και η ομάδα της ΓΚΟΕ ε, μας λέει ότι η κυρία Ρίνα Ρόνια Κάρη θα συμμετέχει στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις επιβεβαιώνεται η ανάλυση των καθηκόντων της. Έχω λάβει ε, προτάσεις από το Συμβούλιο για